Buongiorno, cominciamo anche se un pochino in... Καλημέρα, ξεκινάμε με κάποια καθυστέρηση. Πρώτα έχουμε το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ρωσίας, Ενωσιακός Τελωνιακός Κώδικας μάλλον. Έχουμε πρόταση ψηφίσματος. Η συγγήτης είναι ο κύριος Στέρντι που δυστυχώς δεν είναι εδώ και αντικαθίσταται από τον κύριο Κάμπλ την κυρία, τον κύριο Κάμπολ που παρακαλώ να ξεκινήσει αμέσως την παρουσίαση. Κύριος Βίντερ, Πρόεδρε, αντικαθιστώ εγώ τον κύριο Στόργερ, μου επιτρέπετε. Ελπίζω να μην υπάρχει αντίρρηση. Είχε γίνει κάποια συζήτηση το πρωί. Δεν πάση αντικαθιστώ εγώ τον Ρόμπερτ, λοιπόν. Και αν μου επιτρέπετε να σας εξηγήσω τι θέσεις. Είναι λοιπόν ε, και εισηγητή ε, για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, ο κύριος Στοερδί, ζητεί ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους εδώ παρισταμένους και ιδιαίτερους από εσάς, κυρία Πρόεδρε, που δεν είναι εδώ για να σας παρουσιάσει την ε, σύστασή του. Την γνωμοδότηση λοιπόν θα σας την παρουσιάσω εγώ. Εδώ η Επιτροπή Ίντα εκφράζει συνεχίζει μάλλον στην έκφραση των ελπίδων, των ε, ε, προσδοκιών, των ε, θέσεων της για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, η οποία πρόκειται ύστερα από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων, εφόσον βεβαίως το επικυρώσει η Δούμα, να ενταχθεί στον, στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ε, εκφράζονται οι γενικές ε, προσδοκίες για το τι μπορεί να είναι η θέση της Ρωσίας στο μέλλον, μια ισορροπημένη δηλαδή εμπορική σχέση μεταξύ των δύο μπλοκ και η άρση των αδικαιολόγητων και αθέμητων φραγμών στο εμπόριο για τη δημιουργία ενός μιας αγοράς ελεύθερης και ισότιμης για την κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Όλα αυτά με στόχο να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο εν αναμονή εντωμεταξύ της προφορίας από τη Δούμα. Πιστεύουμε θα έχει εγκρίνει μέχρι το Σεπτέμβριο από πλευράς Ρωσίας. Και έτσι όταν έρθει η ώρα για την επίσκεψη στη Ρωσία θα είμαστε έτοιμοι. Τον Οκτώβριο δηλαδή εφέτος πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στους σκιώδεις εισηγήτες που είναι μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας για τα εμπορικά θέματα για συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία. Η κυρία Βαντέρε για το ΕΛΚ δεν είναι εδώ. Ο κ. Χούτας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Η έκθεση, μάλλον ο εισηγητής, εκπώνησε μια εξαίρετη έκθεση και θα στηρίξει η ομάδα μας την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ, Κόκνε... Κοχμερίν, κυρία Κοχμερίν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Και εγώ αισθάνομαι ικανοποίηση για τα όσα έχει προτείνει ο εισηγητής στο... στην γνωμοδότησή του. και θα ήθελα να αναφέρω κάποιες ε, ερωτήσεις ή ανησυχίες σε σχέση με την μάλλον αισιόδοξη προοπτική και τις ε, προσδοκίες της ε, γεμάτας ελπίδα που ανέφερε ο κύριος Βίνκλερ για τη σχέση με την Ρωσία. Αυτό το λέω διότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας μίλησε, ο Επίτροπος ε, για τις σχέσεις μας ε, με τη Ρωσία, δεν φάνηκε πολύ αισιόδοξο ως προς την ε, σύσφυξη των εμπορικών δεσμών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας μετά την προσχώρηση της Ρωσίας των Ποέτων. αντίον, είπε ο Επίτροπος. Και αυτό δεν το λέει μόνο εκείνος, αλλά και άλλες πηγές. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι αξιοποιούν την προσχώρηση των ΔΟΕ ως επιχείρημα για να μην προχωρήσει σε περαιτέρω απελευθέρωση των ε, εμπορικών συναλλαγών, σε περαιτέρω δηλαδή ε, βελτίωση στις διαπραγματεύσεις και στις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βλέπουμε να έχουμε προχωρήσει αρκετά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καλέσουμε για άλλη μια φορά τη Ρωσία να βελτιώσει τη στάση της, να δείξει πιο θετική στάση. Όλα αυτά νομίζω μπορούμε μέσα στο ψήφισμα να τα ενσωματώσουμε για τις εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία. Γιατί όπως λέμε και στα γερμανικά, κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Ελπίζω να μπορέσουν να με μεταφράσουν οι κοπέλες της καμπίνας. Ευχαριστώ και ο Σούλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον για την προσέγγιση και για τη δουλειά που έκανε και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πολύ καλή συνεργασία στην Νομισματική Επιτροπή για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ρωσία για τις εμπορικές σχέσεις. Να πω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο-τρία σημεία που θα μπορούσα να θίξω όσον αφορά το θέμα για συζήτηση με τον εισηγητή κυρίως στο σημείο 10 του σχεδίου του κειμένου. Ίσως δεν ακολουθεί η σωστή προσέγγιση αν καλούμε να προστατευτούν βασικά στοιχεία. Βεβαίως είναι ουσιαστικά στοιχεία, αλλά φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε σε μια καλή νέα συμφωνία, πραγματικά αξιόπιστη συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία και στον τομέα των εμπορικών σχέσεων. Αν τους θεωρήσουμε ισότιμο εταίρο ο οποίος ενδιαφέρεται για πραγματική συνεργασία και σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει αυτό που συζητήσαμε χθε με τη Δανική Προεδρία, με το πράσινο εμπόριο. Αν δείτε το κεφάλαιο περί ενέργειας, θα έπρεπε αυτό να αναφέρεται εδώ, ότι πρέπει να αναπτύξουμε κοινή προσέγγιση και θέλω να πω ότι ίσως πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης. Πρέπει να ξέρουμε ότι διαπραγματευόμαστε με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να ασχοληθεί με τις δικές της εξωτερικές σχέσεις με τις άλλες χώρες όπως επιθυμεί. Πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς περιγράφοντας τη σχέση με τους εταίρους της Τελωνιακής Ένωσης, με τους άλλους διαπραγματευόμενους εταίρους στην Τελωνιακή Ένωση. Και με τα χαράς να συνεργαστώ περαιτέρω με τον εισηγητή και πιστεύω ότι έχουμε μια καλή, θα έχουμε μια καλή έκθεση στα χέρια μας αργότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μιλήσουν, άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Από πλευρά τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Σημεριζόμαστε απόλυτα τα όσα υπόθηκαν για την ποιότητα της έκθεσης. Είναι πράγματι μια καλή έκθεση. Αλλά θέλω να επανέλθω σε κάτι που ανέφερε κάποιος ευρωβουλευτής και έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε κάπως την εντύπωση ότι η Ρωσία σήμερα θεωρεί ότι ό,τι έχει δώσει στα πλαίσια του ΠΟΕ εμπορικά είναι και το maximum που μπορεί να δώσει. Τώρα είμαστε στο δεύτερο στάδιο που είναι η διαπραγμάτευση της νέας συμφωνίας και έχουμε την αίσθηση ότι δεν θέλουν τίποτα να προσφέρουν. Πια να σας πω και κάτι που ίσως να μην υπάρχει αρκετά σαφώς στην έκθεση και είναι το εξή. Ο πρόεδρος Μπαρόσο το είπε και στον πρόεδρο Πούτιν στην πρόσφατη διάσκεψη ότι για μας δεν θα υπάρξει νέα συμφωνία με τη Ρωσία αν δεν υπάρξει και ένα κεφάλαιο εμπόριο και επενδύσεις που είναι αρκετά ισχυρό και ουσιώδες. Και αυτό είναι ακριβώς που μπλοκάρει σήμερα τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία. Οπότε εγώ αν θέλετε πολιτικά θα τα έβαζα πιο έντονα μέσα στην έκθεση αν εγώ είχα συντάξει την έκθεση αυτή. Δεν είναι κριτική αυτή που κάνω, απλώς ε, σας περνάω έτσι ένα μήνυμα. Και επιβεβαιώνω ότι από πλευρά των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε την αίσθηση ότι τώρα ο ΠΟΕ ε, μπορεί να έχει κάνει ό,τι είχε να κάνει με την Ρωσία, αλλά τώρα πρέπει να υπάρχει και κάποιο αντιστάθμισμα της προσχώρηση των ΠΟΕ. Άρα στον χώρο των επιχειρήσεων, των επενδύσεων με μέτρα τα οποία να μην μπλοκάρουν το εμπόριο. Όλα αυτά που συμβαίνουν όμως τώρα από πλευρά της Ρωσίας είναι ανησυχητικά για μας. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι οι παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη και από τον εισηγητή και από τους ε, συναδέλφους. Στις 25 Ιουνίου το μεσημέρι έχει καθοριστεί η προθεσμία για τις τροπολογίες και θα υπάρξει χρόνος να ε, συζητηθούν αυτά, να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στο σημείο 15, πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, υιοθέτησε η Ολομέλεια στη Σύνοδο ε, του Ινίου ένα ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντερικού Κανονισμού, δηλητώντας από το Συμβούλιο ε, να μην δώσει εντολή για τι διαπραγματεύσει όσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετηθεί για την υποχρεωτική εντολή που ε, προτείνεται. Κατά συνέπεια. Συγγνώμη, αλλά καμιά φορά υπάρχουν κάποια, κάποιες λεπτομέρειες ε, οργανωτικές αποφάσεις αν αποσύρουν οι συντονιστές την πρόταση ψηφίσματος βασιζόμενοι στο άρθρο 90 που ισχύει για την Επιτροπή μας, δοθέντος ότι το ψήφισμα ήδη ψηφίστηκε και οθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του ίδιου κανόνα και για το ίδιο θέμα, ε, ε, ε, επειδή υπάρχει η πρόταση ψηφίσματος αποσύρεται η Επιτροπή μας καλείται να παράγει ένα ψήφισμα για τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή που προτείνεται. Για να μπορούμε να συμβάλλουμε στις εργασίες του Συμβουλίου, πιστεύω ότι η εξέταση του σχεδίου ψηφίσματος θα πρέπει να λάβει χώρα στη συνεδρία σήμαση του Ιουλίου, η ψηφορία στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο και στην Ολομέλεια το αργότερο τον Οκτώβριο. Υπάρχει κάποιος που επιθυμεί να πάρει το λόγο. Καλώς. Πάμε στο σημείο 16, Γενικός προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013. Το επόμενο σημείο είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο. Η συγκεκριτής προσωμοδότηση όσον αφορά τον προπολογισμό ε, είναι ο κ. Στάσνη του ΕΛΚ και το δίνω το λόγο. Αν δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ ο εισηγητής, οπότε ρωτάω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να μας πει. Είναι λίγο μυστηριώδη συνεδρίαση. Άλλο είναι εδώ, άλλο δεν είναι εδώ. Αυτό που είναι εδώ δεν είναι γεγραμμένο να μιλήσει. Αυτό που απουσιάζει είναι γεγραμμένο εδώ για να μιλήσει. Alors, monsieur le rapporteur... Κύριε Σιγητά, όταν είστε έτοιμος, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair, and I apologize. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα κάποιες υποχρεώσεις, βιαζόμουν. Ελπίζω, ότι σε 9.30 θα συζητηθεί το θέμα μου και ακριβώς ε, τώρα συζητείτε, Εγώ φταίω που άρχισα. Να ξεκινήσω ευχαριστώντα την Επιτροπή που θέτει την περσμένη εβδομάδα σαφέστατη γραμμή για εντολή για τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του 2013. Αυτό θα διευκολύνει το έργο μας για το επόμενο βήμα, τη σύνταξη της νομοδότησης για την, τον προπολογισμό και τις ε, τροπολογίες για το σχέδιο προπολογισμού. Οι προτεραιότητε τη Επιτροπή καθορίστηκαν σαφώ στην τελική γνωμοδότηση. Θα ήθελα να παραθέσω τι προτεραιότητε. Η αναθεώρηση τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ενώση για το 2013, κάτι που ζητήσαμε στην έκθεση Κασπαρή για την εμπορευματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώση όσον αφορά τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Ε, υποστήριξη στην διεθνοποίηση των μικροσύνων επιχειρήσεων και μέσω βελτιωμένων κέντρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέσω ε, διαφόρων αγορών και λοιπά που ετοιμάζονται και εκδηλώσεων. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους εμπορικούς εταίρους στη νότια γειτονιά μας ε, σύμφωνα το ότι δίνουν περισσότερα, πάρουν περισσότερα με αυτή την αρχή. Και θέλουμε προπαρασκευαστική δράση για την Ευρωμοσιακή Πρωτοβουλία, για την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε οι και επίσης οι ενισχύσεις για το εμπόριο ICA, ICI Plus να διατηρηθούν και επίση η μακροοικονομική βοήθεια να διατηρηθεί. Πώ εντάσσονται όλα αυτά σε αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο χρόνο, για τον Απρίλιο... Τον Απρίλιο στις 25 του μηνός παρουσίασε το σχέδιο προπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013. Όπως ξέρετε, εν γέννη το σχέδιο προπολογισμού για το 2013 είναι στα 250,9 δις όσον αφορά ανάλυση υποχρεώσεων, 2% αύξηση σε σχέση με πέρσι, ε, λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα πληθωρισμό. Αυτό συνεπάγεται ότι λαμβάνουμε υπόψη τον πληθωρισμό και οπότε ο προπολογισμό παραμένει το ίδιο. Το, το κονδύλι παραμένει ίδιο. Οι πληρωμέ για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 που πρέπει να επανακαταβληθούν πέρσι για το 2013 είναι 137,9 δις, άρα μια αύξηση του 6,8%. Ε, για λεπτομέρειες να αναλύσω την όλη αλλαγή των ποσών που προβλέπονται για κάποια κονδύλια του προπολογισμού στο σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013. Η χρηματοδότηση πολιτού πλαισίου αυξάνεται και για την ανάληψη υποχρεώσεων συν 4,66% για τη χρηματοδότηση συν 22,71%. Αυτό είναι ικανοποιητικό η συνεργασία με τις βιομηχανοποιημένες τρίτες χώρες αυξήθηκε σε ανάληψη υποχρεώσεων κάτω από το επίπεδο του πληθωρισμού, συν 1,58%. Όμως μειώθηκαν οι πληρωμές και αυτό είναι κάπως ανησυχητικό. Είναι το ότι είδαμε μεγάλη αύξηση και σε ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμές για την οικονομική συνεργασία με την Ανατολική Ευρώπη που ευθυγραμμίζεται με τα αιτήματά μας. Δυστυχώς ε, παρατήρησα μια μικρή μείωση μείον 2,73 κατά ανάληψη υποχρεώσεων και 3% στη χρηματοδότηση για το κονδύλι που αφιερωνόταν στην συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας. Ε, και αυτό είναι λίγο προβληματικό διότι η γνωμοδότησή μας τονίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία με εξαγωγικές αγορές που αναπτύσσονται ραγδαίως, αλλά βλέπουμε ότι αυτό αντισταθμίζεται εν μέρη με σημαντικό με συν 59% ανάληψη υποχρεώσεων, σημαντική αύξηση για δραστηριότητε συνεργασία πέρα από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για την Ασία, Κεντρική Ασία και Ιράκ. Και τέλος το κονδύλι για τις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις αυξάνεται κατά 23,3% σε ανάληψη υποχρεώσεων και 18,7% σε πληρωμές. Ε, και εκεί θέλουμε να ευθυγραμμιστεί το πρόγραμμα διαπραγματεύσεων Μάλλον το αίτημά μα να δίνονται περισσότεροι πόροι στα πίστα διαπραγματεύσεων λαμβάνεται υπόψη. Υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Είναι αρκετά λογική η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με της Επιτροπής μας, όμως α, πρέπει σε κάποιους τομείς να γίνουν προσαρμογές για να καλυφθούν οι νέες μας προτάσεις, συνοψίζοντας. Να σας πω τι έγινε στην πρώτη συνεδρία των συντονιστών για τη γνωμοδότηση αφορά τον προπολογισμό τη 9 Μαΐου κατόπιν πρωτοβουλία των Γενικών Συγητών για το, του κυρίου Λαβία, του Γενικού Συγητού για, την, ε, για τον προπολογισμό του 2013. Στη συνάντηση κάλεσε κάθε επιτροπή να καταρτήσει κατάλογο στην γνωμοδότησή του για τομεί που πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια και τομεί όπου θα μπορούσαν να γίνουν περικοπές. θα ήθελα από εσά συνάδελφοι, κάποιες προτάσεις σχετικά και με αυτό το θέμα ε, και προσβλέπω συνεργασία με τους Κιώδης και να ακούσω ποιες είναι οι πρώτες τους ε, αντιδράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως έχει κάποιες προτάσεις, κάτι που θέλει να μας πει. Όχι λοιπόν. Και έτσι στις 11 και 12 Ιουλίου θα εξετάσουμε το σχέδιο. Και τώρα το βλέπετε για τις 10 η ψηφοφορία. Και άρα μας μένουν μερικά λεπτά για να ξεκουραστούμε. Δεκόπτουμε μέχρι τις 10. Υπότιτλοι Bene, Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας εκ νέου. Πρώτα απ' όλα ζητώ από τους συναδέλφους να μου πούν αν συμφωνούν οι διάφορες κάμερες, οι τηλεοπτικές και οι χειριστές τους να παραμείνουν στην αίθουσα να κινηματογραφούν ή αν προτιμούν να βγουν από την αίθουσα, υπενθυμίζοντας όμως τους δημοσιογράφους ότι ένα τέταρτο μετά το τέλος των ψηφοφοριών θα υπάρξει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συνέντευξεων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια αίθουσα που γνωρίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό όσον αφορά την ανακοίνωση στο κοινό, επικοινωνία με το κοινό και το δικαίωμα ενημέρωσης από πλευρά του τύπου υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, ένα τέταρτο μετά ψηφοφορία. Ξέρουμε ότι θα είναι μακρά ψηφοφορία δική μας, θα κρατήσει πολύ. Υπάρχει κάποιο από εσά που επιθυμεί να μην κινηματογραφηθεί, να μην μεταδίδεται η συνεδρίασή μας. Αλλιώς θα αφήσουμε να κινηματογραφούν. καλώ. Δεν υπάρχει αντίρρηση, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τροποποίηση του πρώτου παρατήματος του κανονισμού του Συμβουλίου για να συμπεριληφθούν κάποιες χώρες του καταλόγου των περιφερειών ή των χωρών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Εισηγητής ο κ. David Μάρτιν. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο εκθέσεις που αφορά την νομοθετική αυτή πρόταση που έχει σκοπό να τροποποιήσει τον πρώτο, το πρώτο παράδειγμα του κανονισμού όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Έχουμε τρεις τροπολογίες που κατετέθησαν από την συγκεκριτή, οχτώ από άλλα μέλη και μία από την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 4 και 5 και την ΔΕΒΕ. Είναι ταυτόσιμες τροπολογίες. Υπέρ, υπέρ κατά απορρίπτονται τροπολογία 2 και 6 και αυτές ταυτόσημες εγκρίνονται α συγγνώμη ποιος είναι κατά και ποιος απέχει 7 τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές. Τροπολογίες 10 και 11 και αυτές είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές τροπολογία 3 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Έλεγχος, λέει ο Πρόεδρος. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. accolto, approvato. 32 a favore. 16 accolto, 16 Εγκρίνεται. E Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, διότι υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα και κάποιες κάρτες που δεν λειτουργήσαν. Άρχεται η ψηφοφορία εκ νέου. Il Πέρας. Έχουμε δύο μέλη του ΕΛΚ παραπάνω. Πέρας. 17 υπέρ, 10 κατά, άρα εγκρίνεται. Εμενταμέντο 8. Τροπολογία 8. Υπέρ. Ah, Καταπίπτει. Τροπολογία 5. Ε, ε, ε, τροπολογία 1. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία όσον αφορά την τροποποιηθήσα πρόταση υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Έχουμε έναν ΕΛΚ παραπάνω. Μια ψήφο ΕΛΚ παραπάνω. Μία κάρτα παραπάνω ΕΛΚ έχουμε. Ωρα, Όλα καλά, πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 2 κατά, 9 αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, ξεκινάμε τώρα ψηφοφορία για την νομοθετική αυτή πρόταση. Πέρας. Εγκρίνατε. 25 ψήφοι πέρα, 2 ψήφοι κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Μάρτιν, στον κύριο Μάρτιν. Τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου στον τομέα των εισαγωγών ελαιολάδου και άλλων αγροτικών προϊόντων από την Τουρκία και όσον αφορά τις καταξιζοδότηση ε, πράξεις ε, που θα ανατεθούν στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διάφορες αρμοδιότητες δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι θέμα επιτροπολογίας και τριών κανονισμών. Η συγγετής ο καθηγητής Μορέιρα. Έχουμε τρεις τροπολογίες που αντικατοπτίζουν τις αλλαγές που έγιναν από το Omnibus 1 και Omnibus 2 που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή μας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ δεν κατατέθησαν τροπολογίες. Προτείνω να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες ομαδικά όσον αφορά το σχέδιο εκθέσεως. όλο το πρώτη ομάδα. Μέχρι τη 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογική σκέψη 5, όχι, τελική ψηφοφορία έχουμε λέει πρόεδρος. Όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, καμία ψήφος εναντίον, δύο αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, καμία ψήφος εναντίον μία αποχή εγκρίνεται. Θέλει να διαπραγματευτεί πριν την Ολομέλεια ο ηγητής. Ο κύριος Λάγκε. Όχι. Εκτός μικροφώνου μια απάντηση του κύριου Λάγκε. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Νέας Ζηλανδίας με την οποία τροποποιείται συμφωνία Μηβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Νέας Ζηλανδίας. Ο κύριος ε, Μορέρα είναι συγητής. Δεν υπάρχει κατατεθήσα τροπολογία όσον αφορά το σχέδιο κειμένου. Ψηφίζουμε κατευθείαν την πρόταση με ηλεκτρονική ψηφοφόρια. Άρχεται η ψηφοφόρια. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. 29 ψήφοι υπέρ. Καμία ψήφος εναντίον, καμία αποχή. Συγχαρητήρια ακόμα και αν δεν είναι εδώ κ. Μορέιρα, τροποποίηση της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας. Ο κύριος Μορέιρα είναι ο συγητής. Δεν υπάρχει τροπολογία. Κατατεθήσα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 29 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται τροποποίηση του κανονισμού για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόλιο κρέας υψηλής ποιότητας, το χείριο κρέας, το κρέας των πουλερικών, το σιτάρι και το σιμιγδάλι καθώς και τα πίτουρα και εν γέννη και άλλα υπολείμματα. Στόχος είναι να ο κανονισμός με το καθεστώς μετά αβώνα της κατεξοδότησης πράξης και της εκτελεστικές πράξης. Το σχέδιο έκθεσης έχει πέντε τροπολογίες. για να προσαρμοστεί με την Omnibus 1 και Omnibus 2 που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή μας. Καμία άλλη τροπολογία δεν έχει κατατεθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιήθηκε πέρας ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ. Καμία απόχη, καμία ψήφος. Κατά. Ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ. Δεν έχουμε αποχή, δεν έχουμε ψήφο κατά. Εγκρίνεται. Κύριε Λάγκε, θέλετε κάποιο διάλογο με το Συμβούλιο. Τώρα, μικροοικονομική ενίσχυση προς την δημοκρατία της Κυργυσία. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη δημοκρατία της Κυργυσία. Λοιπόν, θέλει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δοθεί μακροοικονομική συνδρομή στη δημοκρατία της Κυργυσία. Η συγγητής είναι ο Βιτάλ Μορέιρα. Έχουμε μόνο μια τροπολογία για τον εισηγητή. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία που έχουμε τον εισηγητή, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, τέσσερις εποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ. Μία ψήφος εναντίον, τέσσερις εποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ διαπίστωση της συμμόρφωσης και αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων, πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο της προφορικής ερώτησης όσον αφορά τη συμφωνία, όσον αφορά την αξιολόγηση συμμόρφωσης και αποδοχή των μηχανικών προϊόντων για το πρόσθετο πρωτόκολλο ώστε την προφορική ερώτηση να υποβληθεί στην Ολομέλεια του μηνός Ιουλίου. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 27 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, δύο αποχές εγκρίνεται. Θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας. Η κυρία Ζαμόρα είναι η συγγήτρια. Υπάρχουν 23 κατατεθείς ψηφοφορίες για το σχέδιο γνωμοδότησης. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 13, 13 ψήφοι κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 8 και 30 απεσύρθησαν. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσέρισαν οι 31, 9 και 32. Ψηφίζουμε τη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 κατά τμήματα η τροπολογία 33 ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται θα γίνει έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει μια κάρτα ΕΛΚ παραπάνω. Καλώς. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ. 13 ψήφοι κατά. Καμία αποχή απορρίπτεται. Α, όχι, συγγνώμη, εγκρίνεται λέει η Πρόεδρος. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 13 ψήφοι κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, α, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 13 ψήφοι. Κατά καμία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά Α, ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Έλεγχος. Πέραση ψηφοφορίας. Επεκράτησε κάποια σύγχυση. Είδα να σηκώνονται χέρια, αλλά παρόλα αυτά είναι 26, Τέλος πάντων. Κάποιο μπέρδεμα έγινε, ήταν σε κάθε αποτελέσματα. 26-3 εγκρίνεται. Καθυστερεί λίγο η διαρμηνία και γι' αυτό σηκώνται τα χέρια με διαφορετικού ρυθμού. Εντάξει, κανονικό είναι αυτό, συχνά συμβαίνει. Φτάσαμε λοιπόν στην τροπολογία 17 υπέρ, συμβαστική 17 λέει η Πρόεδρος. Πού βρισκόμαστε. 41 στη 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για τον έλεγχο πέρας υπέρ 16 ψήφοι 13 ψήφοι κατά καμία αποχή εγκρίνεται τροπολογία 17 υπέρ κατά ας κάνουμε έναν έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία πέρας 16 υπέρ 12 κατά καμία αποχή εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά Είμαστε στη 18, λέει η Πρόεδρος. 18 υπέρ. Κατά. Να κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 12 ψήφοι κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 καταπίπτει. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Καταπίπτει αν υιοθετηθεί συμβαστική 2, άρα καταπίπτει. Τροπολογία 4 πάμε τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Α, τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται νομίζω, αλλά κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ, δεκατέσσερις ψήφοι κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 28 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 15 ψήφοι υπέρ, 14 ψηφί κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία όσον αφορά την τελική θέση. Πέρας ψηφοφορίας. «22 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 4 απόχες, εγκρίνεται συγχαρητήρια στον συγκητή λοιπόν τροποποίηση της οδηγίας για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας σχετικά με την πληροφόρηση που αφορά εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και της οδηγίας της Επιτροπής. Τελευταία ημερομηνία ήταν η 1η Ιουνίου 2012 για τις τροπολογίες θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά την οδηγία περί διαφανείας. Ο κύριος Χέλμοντ Σούλτς είναι εισηγητής, κατέθεσε τρεις α, τροπολογίες στο ίδιο γνωμοδότης, άλλες τρεις τροπολογίες κατετέθησαν από άλλα μέλη. Θα ακολουθήσουμε τον κατάλογο ψηφορίας και πάμε στο, στην τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 11 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται εκτός αν θέλετε να κάνουμε έλεγχο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Όχι. Να κάνω... Α, κατέπεσε, μην κάνουμε λίγα την 4. Ναι, κατέπεσε η 4. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Στο, όσον αφορά το τροποποιημένο κείμενο. Α, ελέγχουμε το τελευταίο. Την τροπολογία 2. Έλεγχος για την 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 12 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Όσον αφορά τροποποιηθήσα πρόταση, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 26 υπέρ, 2 ψήφοι κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Ετήσιε οικονομικέ καταστάσει, ενοποιημένε οικονομικέ καταστάσει και συναφεί εκθέσει επιχειρήσεων ορισμένων μορφών. Ο κύριο Σούλτ είναι συγητή και έχει υποβάλει 26 τροπολογίε και άλλε 26 κατετέθησαν από άλλα μέλη. Είναι πιο μακρά αυτή, πιο, μεγάλη, πιο μεγάλος ο κατάλογος. Και θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα η Πρόεδρος. Λοιπόν, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία η τροπολογία 1. Πέρας. 15 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται με την ίδια φορά με την προηγούμενη 4 υπέρ, κατά, αποχές θα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την 4. Πέρας. Όπως πριν 15 υπέρ, 14 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας 15 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 και 38 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 5. Πέρας. 16 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 καταπίπτει, διότι εγκρίναμε την 49, άρα δεν ψηφίσουμε. Έτσι λέει εδώ. Ah, 40. Vabbè. Allora, emendamento 15. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία έλεγχος. Ελέγχουμε την τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiuso. Πέραση ψηφοφορία. 15 υπέρ, 14 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 και τροπολογία 41 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνονται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Έλεγχος. Έλεγχος τη 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ. 15 ψήφοι κατά συνεπώς απορρίπτεται καμία αποχή τροπολογία 45 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία έλεγχος Chiuso. Πέρασε τη ψηφοφορία. Κάποιος περισσεύει, έχουμε μια κάρτα παραπάνω. Για ε, κοιτάξτε λίγο, έχουμε έναν παραπανήσιο. Πρόεδρε, ο κύριος Κλάις εδώ είναι από τους μη εγγεγραμμένους. Μας θυμάμαι την παρουσία του, μια σπάνια τιμή και γι' αυτό βλέπετε έναν παραπάνω. Ο κύριος Κλάις είναι. Άρα ψηφίσουν 30 και όχι 29. Από τους μία εγγεγραμμένους ο κύριος Κλάης. Ο Πρόεδρος, χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζω να σας ξαναδούμε. Μας θυμάται και εσείς με την παρουσία σας. Αλλά μετά από αυτή την παρατήρηση έλεγα ότι αν μας είχατε κάνει την παρουσίαση νωρίτερα θα είχαμε κερδίσει και λίγο χρόνο. Ελάτε, ελάτε, αν και δεν επιτρέπετε κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών, εν πάση περιπτώσει, πείτε μας κάτι. Πρόεδρε, εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Πεκάλη και την κυρία Λεπέν που δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες. Και έτσι δεν μπορεί να είναι εδώ. Η Επιτροπή θα πρέπει, έπρεπε να είναι ήδη ενήμερη γιατί ενημερώθηκε χτες μάλιστα κανονικά. Κοιτάξτε, θεωρήσαμε ότι ίσως να υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Σας είχαμε δει πριν. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα όσον αφορά τις ψηφοφορίες ψήφους πάνω κάτω. Έχουμε 15 υπέρ, 15 κατά και γι' αυτό αυτή η τροπολογία τελικά απορρίπτεται. 45 έτσι, υπέρ. Όχι, 46, υπέρ. Παρακαλώ να βλέπω τα χέρια σας. Κάτα. Λοιπόν, να ξανακάνουμε την επαλήθευση <laughs> για να καλομάθουμε και το 30 που δεν το έχουμε συνηθίσει. Άρχη ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Εάν συμφωνεί το ΕΛΚ, δεν γίνεται πολιτεύση. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικός έλεγχος για την συμβιβαστική 7 πέρας της ψηφοφορίας 16 υπέρ 14 κατά χωρίς αποχές εγκρίνεται και έτσι πάμε στην 24 και στην 51 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απόρρεπτεται 26 υπέρ. Κατά Να επαληθεύσουμε την 26. Εντάξει, επαληθεύουμε την 26. Α, τη συμβαστική 8, μάλιστα. Πέρας. 8, άρχεται η ψηφοφορία. πρόεδρε, Δεν υπολογίστηκε η δική μου ψήφος, Πρόεδρε, δεν βλέπω να καταγράφηκε. 15-15 και απορρίπτεται το εκ τούτου. Γιατί αφού είμαστε 30 και έχουν 15 ψηφίσει υπέρ και άλλοι 15 κατά, απορρίπτεται η τροπολογία. Και πάμε στην 26, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ενέα. Ο κύριο Σόλτ, πρόεδρε. Συμβαστική 8 πάλι. Εάν ψήφισαν μόνο 29 και τότε και το αποτέλεσμα ήταν 15 υπέρ και 14 κατά, έχει απορριφθεί. Check, check. Check again αν ε. Ωραία, ξανακάνουμε μια επαλήθευση ηλεκτρονική αν θέλετε εν αυτή περιπτώσει για την συμβιβαστική 8. Il voto è chiuso. Allora, 14 a favore, 7. Πέρας ψηφοφορίας 14 υπέρ, 16 κατά, χωρίς αποχές. Δεν ξανακάνουμε άλλη ψηφοφορία για επαλήθευση, γιατί θα χειροτερεύσει κι άλλο το αποτέλεσμα. Και πάω στη συμβαστική 9 υπέρ. Και κόντρο. Κατά άποχες. Απερίφθη. 10. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ορίστε παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας κατάλογος, ένα λάθος στον κατάλογο μας των ψηφοφοριών και γι' αυτό θέλουμε να απορριφθεί από τους, τα μέλη της ομάδας μας πρώτα σε αυτά. Καλώς. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ψηφοφορία για την 30 υπέρ. Κατά. Πρόεδρε, όχι στην τροπολογία 30, στην τελική ψηφοφορία. Στο σύνολο. Μάλιστα. Ωραία, έχει απορρευ... Έχει εγκριθεί η 30 και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Και πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκαπέντε υπέρ, δεκαέξι κατά και απερίφθη. qualcuno vuole intervenire, do la parola. Εάν θέλει κανείς το λόγο, πείτε μου. Θες να μιλήσεις, κύριος Καζάκ. Πρόεδρε, υπάρχει άλλη μία ψήφος από ό,τι βλέπω. 31 έχουν ψηφίσει τώρα, από ό,τι μας δείχνει ο κατάλογος. We 31, 31 Μα είμαστε 31 στην Επιτροπή μας. Κάποιος έφτασε. Κάποιος κατέφθασε. Alors, petit et moyenne entreprise. Μικρό, μεσές επιχειρήσεις, μικρές και μεσές επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα, ε, εμπορικές προοπτικές, επιχειρηματικές μάλλον προοπτικές. Ησυχία παρακαλώ. Άντε, ένα κουράγιο ακόμα να τελειώσουμε. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού Επί της εκθέσεως πρωτοβουλίας της ΣΥΤΡΑ, ο κ. Γουνκλερνό, εισηγητής, ο συντάκτης, έχουν κατευθεί 55 τροπολογίες, έχουν διατυπωθεί συμβιβαστικές τροπολογίες και ελπίζουμε ότι αυτή η πρόταση θα μπορούσε, θα έχει καλύτερη τύχη από ό,τι είχαμε δει στην προηγούμενη θητεία, γιατί ξέρετε ότι είχαμε την ίδια επιχειρηματολογία και τα ίδια ζητήματα. Αλλά αυτή είναι και η παράδοση στην Ευρώπη. Μιλάμε πολύ, βγάζουμε λίγα αποτελέσματα. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται 2 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται 3 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι περίπλοκη κατάσταση. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Α, έχει καταπέσει 16. Πολύ καλά. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 7 υπέρ, κατά. Υπέρ ή κατά. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ. Επαληθεύουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες... 17 υπέρ 10 κατά 2 αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά ελέγχουμε παρακαλώ Πέρα ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 16 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρασε 18 υπέρ, 13 κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται τροπολογία συμβιβαστική 11 υπέρ. Τι 48? Ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Πρώτα πρέπει να κάνουμε το 48. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και η 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφοφορία για το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότης όπως τοποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 26 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται λοιπόν. Και συγχαρητήρια στον κύριο Βίνκλερ. Θέσπιση ενός μηχανισμού, εταιρική ενός εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Έχουμε λοιπόν πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που θεσπίζει ένα μηχανισμό εταιρική σχέση με τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε και η κυρία Αντρικιένε είναι η συγγητριά μας. Έχουμε 58 τροπολογίες, 35 της συγγήτριας και 23 των άλλων μελών. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχει η Επιτροπή, είναι σύμφωνα με το άρθρο 50, τη συνεργασία. Λοιπόν, τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά σκάμια παλήθευση να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφόρια. πέρα ψηφοφόριας. 18 υπέρ, 12 ψήφοι κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά 43. έλεγχος. Έλεγχος για την 43. Πέρας. Δύο ψήφοι υπέρ. 27 ψήφοι κατά. Αλλά γιατί στο καλό μου ζητήσατε τον έλεγχο. Τέλο πάντων, καταλαβαίνω ότι είναι μια sui generis προεδρία. Είμαι κάπω δύο αριθμοί, αλλά τώρα 27-2 μπορώ να δω τη διαφορά. Ψηφίζουμε τη 44. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Πέραση ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 16 ψήφοι κατά, ε, καμία αποχή απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, το ξανακάνουμε, τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στα παραρτήματα συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά έλεγχος. Γιατί 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 13 ψήφοι κατά, δύο αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 16 κατά, καμία άποχη, απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 6 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. 58 καταπίπτει, όταν καταπίπτει δεν ψηφίζουμε. 58 υπέρ, α κατέπεσε, ωραία ωραία. Τροπολογία 1 στις αιτιολογικές σκέψεις. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 14 ψήφοι κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, Νομίζω καλύτερα να κάνουμε έναν έλεγχο. Ας κάνουμε έναν έλεγχο ακόμα. Πέρας. 24 υπέρ, 7 κατά. Δεν είδα που σηκωνόταν τα χέρια φαίνεται. Πάμε στην τροπολογία 3, 4. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας 15 υπέρ 16 κατά καμία αποχή απορρίπτεται Τροπολογία 15. Υπέρ. Α, 7, 7. Ζητώ συγγνώμη. Αφορά την τελική σκέψη 15. Υπέρ τις 7. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά ας κάνουμε έναν έλεγχο αν και κατά την άποψή μου απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας Όχι, κι όμως με δύο ψήφους πέρασε, εγκρίνεται. 16 υπέρ, 14 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Τροπολογία 11. 10. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. του 24. υπέρ, 4 ψηφίκατα, 2 αποχές, εγκρίνονται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγήτη. Θέσπιση κοινών κανόνων, κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης. νομοθετική πρόταση για κοινού κανόνε, λοιπόν, για διαδικασίε και εφαρμογή μηχανισμών εξωτερική δράση των νόσων που εφαρμόζονται σε κάποια νέα εξωτερικά μέσα που εφαρμόζουν, τα, οδηγούν στην εφαρμογή των μέσων αυτών. Η κυρία Αντρικένε είναι η συγγήτρια. Έχουμε 19 τροπολογίες τη συγγήτρια. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 2 υπέρ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 Ψηφίζουμε ομαδικά τη 13, 14, 15 και τη 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο που τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τα κατάφερα, ναι. Λοιπόν, 23 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Δύο άποχες. Εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Με μηχανισμοί ε, προενταξιακής βοήθειας. Θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση για την πρόταση αυτή που αφορά πρόταση κανονισμού για μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας. Η συγγητής μας είναι ο κύριος Βίνκλερ. Το σχέδιο γνωμοδότηση περιέχει 10 τροπολογίες Λοιπόν, έχουμε τις της τροπολογίας. θα ψηφίσουμε. Τροπολογία 20, υπέρ, κατά, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 18 κατά. 0 αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Καταπίπτει. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 24. Πέρας ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 16 κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 και 25. Είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 26 καταπίπτει, αν δεν κάνω λάθος. Τροπολογία 4 υπέρ. Parce que pas για τη 12, λέει η Πρόεδρος. Πού είναι? Θα ψηφίσουμε την 25. Γιατί οι 2, οι 3 και οι 25 δεν ήταν ε, ταυτόσιμες αλλά συμβατές. Θα έπρεπε να το γράψουμε ότι ψηφίζουμε και τα δύο. Να το έλεγε. Τέλο πάντων δεν το έλεγε. Θέμα γραφειοκρατία, τι να Φυγέ τη γραφειοκρατία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 25 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Όλοι είναι ικανοποιημένοι και αν δεν κάνω λάθος προχωράμε στη 4. Σωστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 είναι συμβατές. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 27. 28 συμβατή και αυτή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο συμβατές, η μία απορρίπτεται και η άλλη εγκρίνεται. Αυτά είναι πράγματα μυστηριώδη στη ζωή. 29 καταπίπτει και αυτό είναι επιτυχία ήδη. 30 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. 8 υπέρ, 23 ψήφοι κατά, 0 αποχές, προφανώς απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος. Ας κάνουμε έλεγχο για την 5. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή απορρίπτεται. Ας κάνουμε έναν ελέγχο. Πέρας. 12 υπέρ, 16 κατά. Δύο αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος πέρας ψηφοφορίας 15 υπέρ 16 κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έτσι φαίνεται. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο? Όχι. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ή απορρίπτεται. απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 λέει η πρόεδρος. Α, 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφοφορία όσον αφορά το τροποποιημένο κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «24 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 4 άποχες, χειροκροτήματα και συγχαρητήρια στον εισηγητή». Και τώρα έχουμε θέσπιση ενός μηχανισμού σταθερότητας. Πρέπει να ψηφίσουμε γνωμοδότηση για νομοθετική εξαφέτηση για την πρόταση κανονισμού που αφορά ένα μηχανισμό σταθερότητας εισηγητής είναι ο κύριος Αμπάντ. Το σχέδιο γνωμοδότηση περιέχει έξι τροπολογίες και κατετέθησαν εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγ, απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος για την εννέα. Απροβάτο. Πέρας. 26 με φοβερή διαφορά. Απόλυτη. Τροπολογία 1 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά α, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 αποσύρθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά απορρίπτεται τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία only 20 voted. Eh, cosa succede? Tutto il mondo ha votato. Avete votato tutti? Si Ψηφίσατε Oli? Πέρας. 24 υπέρ, 4 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Alors, avant de, le, le point 30... Πριν τον σημείο το επόμενο. Ah no, sono ancora indietro, madonna. Allora, le dernier punte della session de vote. Τελευταίο σημείο είναι η εμπορική συμφωνία η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της α, ε, παραποίησης απομίμησης. Ε, το σημείο λοιπόν τη πληροφορία είναι το σχέδιο σύσταση όσον αφορά την έγκριση τη εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση παραποίηση απομίμηση. Ο κύριο Μάρτιν προτείνει η Επιτροπή μα να συστήσει στην Ολομέλεια να απορρίψει τη σύναψη τη συμφωνία. Καταρχάς θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες και μετά το σχέδιο σύσταση. Θα ήθελα να αποσύρω την τροπολογία με παριθμόν 1. Ε, και είναι ταυτόσημη, έτσι. Και, και ταυτόσημη. Ο κύριος Χιέλνερ απέσυρε και την ε, τροπολογία του. Την ένα και τη δύο αποσύρουν. Οι ένα και οι δύο ήδη έχουν αποσυρθεί. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η τροπολογία 3. Εφόσον εγκριθεί, τότε η τελική ψηφοφορία για το σχέδιο σύστασης αναβάλλεται μέχρι να έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν απορριφθεί, τότε τελική ψηφοφορία για το σχέδιο συστάσεων του εισηγητή η αρχική. Για το σχέδιο σύσταση την αρχική του εισηγητή. Ναι, η αρχική, δεν είναι αρχικός εισηγητής, η σύστασή του είναι. Συνεπώς ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία αριθμός 3. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. 13 υπέρ, 19 κατά.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 Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Γιατί είχαμε μια μυστηριώδη ψήφο. Λοιπόν, ψηφίζουμε και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορία. Εντάξει. Ωραία το μηχάνημα περιμένουμε να καταλάβει ότι τελείωσε. Α, το κατάλαβε και μας δείχνει τα αποτελέσματα. Ε, έχει καλώς. Συνεπώς, 12 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε η τροπολογία, έτσι δεν είναι. Τώρα. Η πρόεδρος μιλάει με τη γραμματεία. Ε, parce que si c'est adopté, la recommandation est de rejeter Et si ce vote est rejeté, la recommandation d'INTA est donnée approbation. Donc c'est un peu contre. Ε, σκουζάτε, εκεί per chi aveva studiato. Συγγνώμη, για όσους μελέτησαν την ελληνική φιλοσοφία, αυτό είναι κάτι που θέλει, φαίνεται ερετικό και σημαίνει και το αντίθετο από αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, σας διαβάζω. Είσαστε πιο ευφυείς από μένα και λέτε ότι με αυτό που σα διαβάζω εσεί θα καταλάβετε τα πάντα. Και εγώ είμαι βέβαια θα καταλάβετε. Διαβάζω λοιπόν. Είπα... Εάν απορριφθεί η τροπολογία 3, τότε τελική ψηφοφορία για το σχέδιο σύσταση του αρχικού εισηγητή, σα τα είπα και πριν αυτά. Αν εγκριθεί, όπω έγινε στην περίπτωσή μα, τότε σύσταση τη ΣΥΝΤΑ στο Κοινοβούλιο είναι να απορρίψει την άκτα. Αν απορριφθεί η σύσταση τη ΣΥΝΤΑ στο Κοινοβούλιο, στην περίπτωση ισοψηφία, τότε απορρίπτεται το αποτέλεσμα. Για να τα ξέρετε όλα αυτά. Τα ξέρατε και πριν. Ωραία, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Πέρα στις φοφορίες και έχουμε τα αποτελέσματα. Abbiamo 19 a favore. 19 υπέρ, 12 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Παρακαλώ οι δημοσιογράφοι να βγουν από την αίθουσα. Θα υπάρξει συνέντευξη τύπου σε ένα τέταρτο. Και παρακαλώ τους ε, συναδέλφους να να ζητήσουν και από τους δημοσιογράφους να, να κάνουν αυτό που είπα. Να βοηθήσουν να φύγουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Για τους δημοσιογράφους σας είπα, σε 15 λεπτά έχουμε συνέντευξη τύπου. Πηγαίνετε στην ε, συνέντευξη τύπου παρακαλώ. Καλά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 Αλλά αν δεν φοράτε ακουστικά, πού να καταλάβετε τι λέω. Καθίστε στη θέση σας. Διότι δεν τελειώσαμε, δεν τελείωσε η συνεδρίαση. Αν θέλετε να πάτε συνέντευξη τύπου, πηγαίνετε γρήγορα, χωρίς να μιλάτε. Διότι εδώ πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.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 να καθίσουν, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Peut-être que sera mieux, de, faire suspension. Bene, riprendiamo. Καλώ συνεχίζουμε τις εργασίες μας για τους ελάχιστους που παρέμειναν ως ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, μια στρατηγική για την ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Στις 8 Φεβρουαρίου η Επιτροπή ΙΝΤΑ ε, οργάνωσε με την ΑΦΕΤ μαζί ένα εργαστήριο όσον αφορά τη στρατηγική τη ψηφιακή ελευθερία και την ασφάλεια ψηφιακή όσον αφορά την εξωτερική πολιτική τη Ένωση και το ρόλο των επιχειρήσεων. Αυτό το εργαστήριο ε, ξεκίνησε μια σειρά τεσσάρων εργαστηρίων που διοργανώθηκαν σε αφορά το θέμα του διαδικτύου. Η κυρία Ζάξ Τρισάλτε αναθεώνει μια έκθεση όσον αφορά τη στρατηγική της ψηφιακή ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης για την ΑΦΕΤ, η της για γνωμοδότηση είναι η Αμέλια Άντερς Ντότερ. Και τώρα θα κάνουμε πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ζητώ από την κυρία Anders Dotter, την εισηγήτριά μας, ε, αν θέλει να μας πει κάποια πράγματα για το θέμα. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα αυτό. Θέλω να αναφερθώ στην ε, πρωτοβουλία της κυρίας ε, Σχάκε της Επιτροπής για τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Επικεντρώνεται στην στρατηγική μας για τα ψηφιακά δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή μας, ίντα, πολλές φορές κάνει ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τρίτες χώρες. Η κυρία Σχάκε, λοιπόν, θέλει να συμπεριλάβει και αυτή την εμπορική πτυχή Από τις συζητήσεις μας γνωρίζουμε ότι οι εμπορικές σχέσεις επηρεάζουν πολύ την κατάσταση στις τρίτες χώρες. Οι νέες τεχνολογίες ε, όντως επηρεάζουν πολύ την κατάσταση. Πρέπει να δούμε πώς εμφανίζεται ένας εμπορικός χώρος, τι διευκολύνσεις υπάρχουν μέσω του διαδικτύου, τι πληροφορίες παίρνουν οι ίδιοι πολίτες μιας χώρας κλπ. Πέρυσι είχαμε ένα νέο παράδειγμα για τις νέες υπηρεσίες του διαδικτύου και πώς αυτές ανοίγουν νέες δυνατότητες. Όχι μόνο έκφρασης των πολιτών, αλλά ακόμα δίνει το διαδίκτυο και τη δυνατότητα να πέσουν κυβερνήσεις. Συνεπώς, γι' αυτό ακριβώς και εγώ λέω ότι τα δικαιώματα σε κάποιο είδους υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν την πρόσβαση στην ενημέρωση των πολιτών. Άρα και την ενημέρωσή τους για τις αγορές. Είναι προφανές ότι σε πολλές χώρες δεν εφαρμόζονται εξαιρέσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των δημιουργών, γιατί η ψηφική μας ατζέντα μας προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών. Αυτό το θέμα Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες και θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέρφους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρίσταται. Είναι εδώ. Η Σκιώδης. Η συγγήτρια. Παρακαλώ. Thank you, um, Σχάκη. Ευχαριστώ πολύ δεν είμαι μόνο σκιώδης εισηγήτρια στην ίντε, αλλά είμαι και εισηγήτρια στην Επιτροπή ε, Επιτροπής Γι' αυτό και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Έχω ζητήσει και από τους σκιώδεις και από οποιοδήποτε άλλο ευρωβουλευτή, ακόμα από τις επιχειρήσεις ή από την κοινωνία των πολιτών, όποιο θέλει να σχολιάσει να το κάνει. Γιατί όντω είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει την καθημερινή ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Προς το παρόν είμαι εδώ για να ακούσω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Εκτός μικροφώνου η πρόεδρος, δυστυχώς δεν ακούμε. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκλωριόζο, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Για την κυρία Σάκε θα ήθελα να πω απλώς ότι είμαστε εδώ για να την ακούσουμε, για να παρακολουθήσουμε την, ε, τις εξελίξεις στην εκθεσή της. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και κάποιο καιρό έχει παρακολουθήσει το θέμα αυτό με τη στρατηγική της που στόχο έχει να βελτιώσει τις στρατηγικές της επικοινωνίας και να τις αξιοποιήσει για την προαγωγή των ανθρωπινών δικαιωμάτων και την προστασία τους. Μπορώ ε, να ακούσω τις ερωτήσεις και να δώσω απαντήσεις, δεν χρειάζεται όμως νομίζω τώρα να δώσω λεπτομέρειες για το σχέδιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Vous voulez... Euh, Ευχαριστώ. Θέλετε, όχι. Δεν θέλει κάτι άλλο να επανέλθει. Και ως εκ τούτου έχουμε την κυρία Σάκε, συγκέντρια. Κύριε Άντερ Σότερ. Το χρονοδιάγραμμα είναι 19 Ιουνίου 19, 20, 19 Ιουνίου είναι η ΑΦΕΤ. Είναι 20 και 21 Ιουνίου, 11-12 Ιουλίου, συναντήσεις, 19 Ιουλίου προθεσμία υποβολής τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι έγκριση στην Επιτροπή προβλέπεται στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Η ΑΦΕΤ όμως θα ψηφίσει στις 20. Θα συζητήσει τουλάχιστον στις 20 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Περνάμε σε άλλο θέμα. Προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακου. Εγώ είμαι η συγγήτρια Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό στην της Ευρωπαϊκή Ένωση στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Βάμβακο. Είναι μια, ένας προσπάνιος ε, διεθνής α, φορείς σε αυτό το τομέα που δεν είμαστε μέλος. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητήθηκε για να δώσει την έγκρισή του όσον αφορά την προσχώρησή μας αυτή. Στη προηγούμενη συνεδρίασή μας θα θυμόσαστε ότι είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με διάφορες πλευρές. Εξετάσαμε το θέμα αυτό και είδαμε και τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα πρέπει να συζητήσουμε τα υπέρ και τα κατά της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή. Είναι σίγουρα ένα θέμα σημαντικό αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους περιορισμούς, την αναπτυξιακή αραιογή, τους δασμούς, την παιδική εργασία κλπ. Μια που είμαι συγκήτρια, πρέπει να είμαι και σύντομη. Αλλά θέλω να πω ξεκάθαρα τη γνώμη μου. Όπως ξέρετε, η ΚΑΚ έχει ως στόχο να συγκεντρώνει τις χώρες παραγωγούς βάμβακος για να διασφαλίζει τη διαφάνεια στην παγκόσμια αγορά του προϊόντος αυτού. Για τη συγκομιδή, για τα στατιστικά στοιχεία, για την οικονομία κτλ. Σε αυτό το συμβούλιο συμμετέχουν η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Φιλανδία, που στις 31 Ιουνίου λίγη η θητεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μπει σαν μια χώρα δυνάμει το άθου 207 της συνθήκης της Λισαβόνας. Πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα συνδέεται με τις λεπτομέρειες. Δηλαδή σε αυτή την οργάνωση, ίσως που είναι η μοναδική στον κόσμο τώρα πια, ψηφίζουν μια ψήφος κατά κεφαλή που για κάποιους φορείς Σίγουρα είναι παλιά μέθοδος, αλλά ακόμα χρησιμοποιείται και επίκαιρα σε οργανισμούς όπου βλέπουν να συμμετέχουν εντός τους σαν ενιαία εκπροσώπηση διάφοροι οργανισμοί που απαρτίζονται από περισσότερες συνιστώσεις, προφανώς αυτό δημιουργεί προβλήματα και δύσκολο κυρίως όταν μετά ε, υπάρχει μια εκπροσώπηση διαφορετικά, διαφορετική από την έποψη του αριθμητικού βάρους κάποιων χωρών σε συγκρίση με άλλες. Όπως γνωρίζετε, ε, εμείς είχαμε υιοθετήσει την ψηφοφορία τη σταθμισμένη κλπ. κλπ. Γι' αυτό η είσοδο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως εντός αυτού του Συμβουλίου ε, είναι σίγουρα ένα έξοχο σήμα, μήνυμα όχι μόνο για καλύτερη διοργάνωση των κεκτημένων μας ή των αγορών μας και των πωλήσεών μας στον τομέα αλλά για να δείξουμε και μια παρουσίαση ε, να έχουμε παρουσία με καλύτερο έλεγχο. Διότι είχαμε το, το πρόβλημα που μας απασχολεί τα παιδιά που εργάζονται αντί να πάνε στο σχολείο ή για κακούς κοινωνικούς κανόνες που ισχύουν για τους εργαζομένους σε κάποιες χώρες σε αυτό το τομέα ακριβώς. Αλλά τούτων λεχθέντων, δηλαδή πότε θα, τι ήταν, πότε θα ήταν χρήσιμο και τι είναι χρήσιμο για μας θα πρέπει να πούμε μεν ότι υπάρχει και ο ύφαλος της ψηφοφορίας. Η Ευρώπη που σήμερα έχει 8 χώρες που εκπροσωπούνται, άρα μετρά 8 ψήφους, θα βρεθεί αύριο να έχει μία ψήφο. Και αυτό ε, θα ήταν επιζήμιο και για τις 8 χώρες που είναι παρούσες και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μαζί με την Ένωση θα έμπαιναν συμμετέχουσες στην, ε, στον οργανισμό αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε, να το εξετάσουμε το θέμα και να υποβάλουμε τροπολογίες οι οποίες να είναι κατάλληλες ε, για την επίλυση του προβλήματος. Υπάρχει και ένα οικονομικό πρόβλημα που είναι της ποσοστώσεως που θα πρέπει να διτεθεί. Η Ένωση ε, θα πρέπει να πληρώσει τις εισφορές ε, και θα πρέπει να πληρώνει και έξτρα ε, συνεισφορά για τη στάθμιση. Και θα δημιουργήσει, αν γίνει κάτι τέτοιο, κακό προηγούμενο, στο οποίο θα μπορούσαν να προσφύγουν και άλλοι οργανισμοί παρομοίου τύπου ε, που αντιμετωπίζουν κρίση όσον αφορά τα οικονομικά τους. Γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε διαφορετική ρύθμιση αφορά την ψηφοφορία και δεύτερον, να υπάρχει διαφορετικό κόστος οικονομικό για την είσοδο μας σε αυτό τον φορέα θα πρέπει να έχουμε μια εισφορά ε, ενία όπως τα άλλα μέλη ή μια αντισταθμιστική ε, εισφορά στα πλαίσια που θα μπει, θα εφαρμοστεί σταθμισμένη ε, ψηφοφορία που θα αναγνωρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει μορφή όπως έχει στη συμμετοχή της άλλους οργανισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για λόγους συντομίας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους ε, που είναι παρόντες και ζήτησαν το λόγο και πρώτα απ' όλα στον κύριο Κούτας. Chair. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό να γίνουμε μέλος της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής, ε, αλλά και πάνω απ' όλα ε, παρακολούθηση της πτυτικότητας των τιμών, της παραγωγικότητας, αλλά και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Πρόκειται για στόχους πολύ σημαντικούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προσχώρηση λοιπόν στο Εθνικό αυτό οργανισμό, στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος, την ΙΚΑΚ, θα έχουμε λόγο σε πολύ σημαντικά θέματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω, θα έχει σημαντική επίδραση, επιρροή και στο θεματολόγιο που απασχολεί την ε, Συμβουλευτική Επιτροπή. Θα επικοινωνούμε επίσης με χώρες ε, παραγωγούς όπως το Ουσμπεκιστάν και άλλες που αναφέρατε, με προβλήματα όπως αυτό της καταναγκαστικής εργασίας των παιδιών που επισημάνατε και εσείς. Όπως είπα, χαίρομαι ιδιαίτερως που δεχθήκατε τη σύστασή μου από την έκθεση για το εμπόριο κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουσπεκιστάν, όπου ζητούμε να παρακολουθείτε καλύτερα η τήρηση των αρχών του εμπορίου και της παραγωγής στην αλυσίδα της παραγωγής. Ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Όπως είπα, είμαι πεπισμένος ότι η έκθεση μας θα υποστηρίξει πλήρως την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Κούτας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε στο ε, στην εργασία των παιδιών και στον τομέα του βάμβακου αλλά και σε κάθε άλλο τομέα. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί και κάνουμε εναντί κάθε κράτους εμπλεκομένου τη μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι και ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος στην υπόθεση αυτή. Η κυρία Κέλλερ έχει ζητήσει το λόγο, αν δεν κάνω λάθος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το έγγραφο εργασία. Έχω κάποιες ερωτήσεις μόνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάς και η ε, Ισπανία μόνο παράγουν ακόμη ε, βάμβακα, αλλά με τίμημα πολύ σημαντικές επιδοτήσεις στους παραγωγούς θα ήθελα να ρωτήσω αν συνεχίζεται αυτό. Και επίση η Ελλάδα και η Ισπανία είναι επίση μέλη τη ΙΚΑΚ, τη Διεθνού Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακο. Ρωτώ λοιπόν πώ θα μπορέσει η εκπροσώπηση της, η αντιπροσωπεία μάλλον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εκπροσωπεί την Ένωση, πώ θα διαφυλάξει και τα συμφέροντα τη Ελλάδα και τη Ισπανία εφόσον προσχωρήσουμε. Επίση, αναφέρεται στο έγγραφο η καταπολέμηση των επιδοτήσεων και των περιορισμών εξαγωγών. Στο ίδιο κεφάλαιο στο σχέδιό σας γιατί αντιμετωπίζετε τα δύο αυτά θέματα από κοινού και γιατί θεωρείτε ότι μπορούν ε, οι περιορισμοί εξαγωγών να οδηγήσουν κάποιες χώρες στην διαφοροποίηση σε πιο ε, μεγάλης προσθεμένης αξίας παραγωγή, όπως λέτε. Επίσης, το θέμα της πτυτικότητας των τιμών που αναφέρατε. Δεν λέγεται τίποτα για την ε, αυξανόμενη τελειοποίηση της αγοράς βάμβακος που την καθιστά πιο ε, την εκθέτει περισσότερο, δηλαδή στην, ε, την καθιστά πιο ευάλωτη στην ποιοτικότητα των τιμών. Σε αυτό δεν λέτε τίποτα. Και κάτι τελευταίο όπου αναφέρεται, αναφέρεστε στις ευρωπαϊκές συμφωνίες θερικής σχέσης της ΕΕ με τις χώρες παραγωγούς το Μπενίν, τον Μπάλι, το και να Φάσο, το Τσάτ, ταυτόχρονα και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και άρα έχουν ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς δηλαδή δασμούς, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι, Συμφωνίε οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, εμπορικές, ιστορίες, ε, εμπορικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Τι άλλο θα προσθέσουν για τις χώρες αυτές, τι θα τους προσφέρουν. Ευχαριστώ, Κέις. Επιτροπή. Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να πω ξεκινώντας ότι είναι ευπρόσδεκτη η έκθεση της κυρίας Μουσκαρτίνη. Υποστηρίζουμε βέβαια την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΆΙΚΑΚ. Οι παρατηρήσει τη κυρίας Μουσκαρντή είναι ακριβώς, είναι ταυτόσιμες με τα θέματα που μας απασχολούν και εμάς και τι έχουμε συζητήσει και στο Συμβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν ένα σχέδιο απόφασης για ένταξη στην ΆΙΚΑΚ, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή στα ε, δικαιώματα ψήφου και στις συνεισφορές θα πρέπει να μας απασχολήσουν περαιτέρω. Θα τα συστήσουμε λοιπόν κι άλλο. Ε, προτείνουμε ως ένα μέλος και με μία ψήφο, με μία μόνο συνεισφορά δηλαδή, να ενταχθούμε. Το θέμα όμως ε, που τοποθετήθηκε ως προς τον περιορισμό της επιρροής, γιατί τώρα έχουμε 7-8 διαφορετικές ψήφους και μετά θα περιοριστούμε σε μία μόνο, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ίσως θα πρέπει να το δούμε μετά την ένταξή μας, γιατί όπως υπόθηκε το καθεστώς ε, που ισχύει στις ψηφοφορίες είναι από τα πλέον ε, παλαιά. Είχε ξεκινήσει δηλαδή με το Κοινό Συμβούλιο Βασικών Αγαθών ε, και ίσως ε, αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια προσπάθεια να το τροποποιήσουμε άπαξ και μετατραπούμε σε μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης, μια ερώτηση σχετική με την προστασία των συμφερόντων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι παραγωγή Κοιτάξτε να σας πω. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό ακόμη και από άλλες ε, σχέσεις, επικοινωνία. Δηλαδή, πριν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπήσει, πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ζητεί από το Συμβούλιο να διαμορφώσει μια κοινή θέση για τα θέματα που υπάρχουν στη μέση διάταξη και έτσι μπορούν τα κράτη-μέλη να επισημάνουν ζητήματα που θα ήθελαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει κατά τη συνεδρία ε, της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής και πιστεύω ότι έτσι λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστημα επιπλέον. Τα κράτη-μέλη τα οποία όλα τα κράτη-μέλη για την ακρίβεια μπορούν και αυτά να μας ε, συνοδεύσουν, να μας ακολουθήσουν στις συνεδριάσεις του ε, Τη συμβουλευτική επιτροπή. Επομένω, ε, πάντα σε κάποια τέτοια Συμβουλευτική Επιτροπή, κράτη-μέλη τα οποία έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα παρίστανται και ενημερώνονται εγκαίρω και συζητούν βέβαια και τα θέματα σε πρώιμο στάδιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, το θέμα της εργασίας των παιδιών και άλλε κοινωνικέ διατάξει μα απασχολεί ιδιαίτερω. Ελπίζουμε ότι με την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μιλάμε με, με, μία φωνή θα έχουμε μεγαλύτερη επιρροή στα θέματα αυτά. Υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση και τη σύσταση. Και η σύστασή μας θα ήταν να πραγματοποιηθεί η προσχώρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως και τους συναδέλφους που μίλησαν. Ίσως να μην ήμουν αρκετά ξεκάθαρη εγώ στην, στο κείμενο που διανεμήθη ή στην παρουσίαση που έκανα σήμερα το πρωί. Επαναλαμβάνω ότι πιστεύω σημαντικότατη την προσχώρησή μας, αλλά πιστεύω σημαντικότατη την ένταξή μας εάν έχουμε ένα σύστημα ψηφοφορίας διαφορετικό, διότι στην Επιτροπή Όπω λέει και μια παροιμία υπάρχει σε πολλές όταν περάσει η γιορτή ε, τελείωσαν όλα. Δηλαδή, ε, οι διαπραγματεύσεις ε, γίνονται πλέον πολύ πιο δύσκολες, γιατί παρετούμεθα από 8 ψήφους για να έχουμε μία. θέλουμε τελικά να μπούμε με, σε, με, με ψηφοφορία που πηγαίνει προς την κατεύθυνση που ε, θέλουμε. Σήμερα έχουμε 8 ψήφους που προστατεύουν τα σύνορά μας και μετά θα έχουμε τίποτα. Διότι θα μετράμε μόνο με μια ψήφο όταν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον τα συμφέροντά μας είναι και συμφέροντα οικονομικά αλλά έχουμε και συμφέροντα διοντολογικά, ηθικά για την προστασία των παιδιών, για τα δικαιώματα των παιδιών, για την ε, προστασία του περιβάλλοντος που πρέπει να είναι μια κοινή δέσμευση. Ε, δεν μπορούμε να πάμε και να, ε, να διαπραγματευτούμε μετά. Πρέπει πριν να διαπραγματευτούμε, διότι διαφορετικά μπορούμε να πούμε μας μείνουμε όπως είμαστε και σας ασκήσουμε πιέσεις Ω σαν Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Όπως το κάναμε σε κάποιες άλλε ευκαιρίες. Λοιπόν, είναι με τη συνένεση των συναδέλφων. Δεν χρησιμοποιώ πληθυντικό βασιλικό όταν χρησιμοποιώ πληθυντικό. Λέω ότι μιλάμε μαζί γιατί είμαστε μαζί. Θέλουμε, επιθυμούμε αυτή τη συμφωνία. Είναι σημαντική συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να γίνει όταν θα υπάρξει πρώτα ένα σύστημα ψηφορίας που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του οργανισμού αυτού να πετυχαίνει τους στόχους της και τους εμπορικούς και τους κοινωνικούς. Νομίζω ότι έτσι απαντώ και στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των συναδέλφων που ακούστηκαν πρώτα. Τώρα εμείς θα τα ξαναπούμε τον Ιούλιο 11 και 12 Ιουλίου για να ξανασυνομιλήσουμε αυτό το θέμα. Στις 13 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία την υποβολή των τροπολογιών. Η έκθεση θα ψηφιστεί 17-18 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να πάει στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσω ότι οι σκιώδεις συγητές είναι ο κύριος Κούτας, Κατζάκα, Καμάλ, Τώρα αν υπάρχουν και άλλοι δεν ξέρω που θα προσθεθούν. Όσον αφορά αυτό το θέμα συζητήσαμε αρκετά το ζήτημα αυτό. Πάμε τώρα. Α, συγγνώμη, ορίστε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πρότεινα ένα ψήφισμα και είχα καταλάβει ότι συμφωνούσατε. Δεν βλέπω να είμαστε πολύ βέβαια εδώ, αλλά ίσως θα πρέπει να δούμε αν συμφωνούν και οι συνάδελφοι και αν μπορούμε τελικά να ετοιμάσουμε ένα τέτοιο ψήφισμα. Βέβαια, βέβαια. Χθε το έγραψα, δεν ξέρω αν κατέφτασε η επιστολή. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που εξέφρασαν σύμφωνη άποψη με αυτά που είπαμε πριν και μπορεί να ενδιαφέρονται, εγώ θα έλεγα να ετοιμάσετε εσείς ένα κείμενο που να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε όλοι μαζί, ούτω ώστε να έχουμε ένα κοινό κείμενο που να το υποστηρίζει όλη η Επιτροπή. Τέλεια. Υπάρχουν άλλοι που το λόγο. Όχι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε τον τελωνιακό κώδικα της Ένωσης. Είμαι πάντα εγώ εισηγήτρια και για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δημιουργεί ένα τελωνιακό κώδικα της Ένωσης. Αυτή η πρόταση της μεταρρύθμισης αναδιατύπωσης που προτείνεται θα επικαιροποιήσει τον κανονισμό για τον εξυγχρονισμό του κώδικα να συνάδει και με την στατική που ακολουθείται μετά την Λισαβόνα αλλάζοντα τον κώδικα τη Ένωση, τον τελωνιακό, αλλά και όσον αφορά την, την ανάθεση εξουσιών. Η, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Εσωτερικού Εμπορίου έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή και εσείς πρέπει επίση να κάνετε τα σχόλιά σα. Είμαι συντάκτρια γνωμοδότησης. Θα συζητήσουμε και με τους παρόντες εδώ, αλλά πρώτα θα πάρω εγώ το λόγο ο η κυρία Κωνσταμερίν και η κυρία Κλάκεν. Είναι σκιώδεις συζητητές. Α, και την Επιτροπή θα ακούσουμε βέβαια μετά. Το σχέδιο κανονισμού το οποίο εξετάζουμε. Κατά τη σειρά ετών τροποποιήθηκε πολύ, υιοθετήθηκε το 2008 όπως γνωρίζετε και ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Εν τω μεταξύ όμως έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνα. Η Ένωση άλλαξε τις λεπτομέρειες συμμετοχής των κρατών μελών και των διαφόρων φορέων στις διαδικασίες. Αλλάζοντας διάφορες διαδικασίες στην επεξεργασία των κανονισμών που συζητούμε, μιλάμε για εκτελεστικές πράξεις ή κατεξουσιδότηση πράξεις. Άρα είναι θεμελιώδες να επανεξετάσουμε υπό το φως των διατάξεων που απέρασαν από τη Λισαβόνα το κείμενο του νέου κώδικα για τα τελωνία που θα πρέπει να απλουστευθεί και θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2020. Γνωρίζετε ότι μετά θα υπάρξει κάποια περίοδος, πώς να το πω, έντασης, διότι ο παλιός κώδικας που ετέθη σε ισχύ, που εγκρίθηκε μάλλον, αλλά δεν ετέθη σε ισχύ, εκεί ανέφερε διάφορους όρους που, για πριν το 2020 για να εφαρμοστεί και ο νέος κώδικας, όμως εντωμεταξύ ε, χρειάζονται ελάχιστες προδιαγραφές που εξακαθαρίστούν, αλλιώς δεν θα το πετύχουμε. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά μόνο την έλλειψη εναρμόνισης και περιοριστικούς όρους σε σχέση με το κείμενο του 2008, αλλά και χρήση κατεξοδότηση πράξης σε κάποιες περιστάσεις που είναι απαραίτητο για ταχεία απλούστευση του κράτους. Μέχρι το 2020 όσον αφορά το σύστημα το το ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να σωματωθεί σε ρυθμιστικό κείμενο, ε, που θα επόκειται σε εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά την αναγνώριση διαφόρων συμφωνιών, το θέμα των μη προτιμησιακών κανόνων προέλευση για τα εμπορεύματα που έρχονται από τρίτε χώρε, για την αξία που έχουν στα τελωνία και όσον αφορά τι σχετικέ δομ που οφείλονται σε ε, διάφορες παρεμβάσεις, ιδιωτικές ασφαλίσεις κλπ. και διαδικασίες που δεν είναι ξεκάθαρες. Και το λέω απευθυνόμενοι τώρα αυτό που λέω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι εμείς θα κάνουμε δουλειά καλή ή θα χάσουμε χρόνο διαφορετικά. Το Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Σύστημα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί διότι είναι προφανές ότι δεν ε, χρειάζεται το εσωτερικό αυτό αλλά αφορά το, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες, όχι το εσωτερικό που αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και το θέμα του χρόνου του ανοίγματος του συστήματος. Και το θέμα πόσε ώρε μένουν ανοιχτά τα τελωνία. Υπάρχουν τελωνία που παραμένουν ανοιχτά περισσότερο, ανοιχτά και άλλα τελωνία λιγότερο. Υπάρχουν ήδη ελέγχου, πιο αυστηρή έλεγχη σε κάποιε χώρε και σε κάποια λιμάνια κάποιων χωρών. Άρα ήδη σε μια χώρα, στην ίδια τη χώρα, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να εφαρμοστούν οι έλεγχοι. Και πάνω απ' όλα υπάρχουν διαφορετικοί έλεγχοι από χώρα σε χώρα στα τελωνία. Και αν προσθέσουμε σε αυτό ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα σύστημα φορολογικό εναρμονισμένο, Έχουμε παραδείγματο χάρη χώρες που εφαρμόζουν το 19% ΦΠΑ, χώρες που εφαρμόζουν το 21% ΦΠΑ. Με αποτέλεσμα προφανές ότι τα περισσότερα εμπορεύματα που εισέρχονται πάνε εκεί που πληρώνεται χαμηλότερο ΦΠΑ. Είναι προφανές και πληρώνοντα χαμηλότερο ΦΠΑ πηγαίνοντας σε άλλη χώρα σε αυτή τη χώρα όπου τα εμπορεύματα εκτολονίζονται, υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα για τον τομέα των μεταφορών μεταφορών εμπορευμάτων προς άλλες χώρες. Γι' αυτό η εναρμόνιση των τελωνίων για μας ε, σημαίνει εναρμόνιση των συστημάτων των ελέγχων, εναρμόνιση των διαδικασιών και εναρμόνιση των συστημάτων των πληρωμών. Διότι όταν παραδείγματο χάρη, δεν ξέρω αν το ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τις διάφορες επιστολές και ερωτήσεις που έχουν τεθεί, έχω στείλει επί το θέματος, με ελάχιστη ικανοποίηση στον φάτσα απαντήσεις, διότι στην Ιταλία υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο ο εισηγητής, αυτός ο φορέας που εισάγει, πληρώνει σε κάποιον εκτελονιστή χρήματα που θα είναι το κόστος του ΦΠΑ, το κόστος εισαγωγής. Ο εκτελονιστής έχει την υποχρέωση για να έχει δικαίωμα να κάνει αυτή τη δουλειά να έχει ε, ασφάλιση. Μετά, όπως συχνά δυστυχώς συμβαίνει, Λίγο συμβαίνει, αλλά συνέβη τέλο πάντων και συνέβη και σοβαρό γεγονός, Διεφθαρμένο τώρα εκτελονιστή που πήρε χρήματα από τον εισαγωγέα, αντί να πληρώσει το τελωνίο, τσεπώνει τα χρήματα και την κάνει. Τι συμβαίνει, ότι η ασφάλεια με την οποία να έχει ασφαλιστεί πληρώνει το τελωνίο. Εν αυτή περιπτώσει το Ιταλικό κράτος αλλά ο εισαγωγέας που την πάτησε θα πρέπει να ξαναπληρώσει την ασφάλιση. Οπότε ε, έχουμε τη μοναδική περίπτωση στον κόσμο όπου μια σύμβαση μεταξύ δύο ατόμων επηρεάζει έναν τρίτο ε, εν αγνία της συμβάσεως και λήψη ευθύνης του. Θα μου πείτε ότι ονειρεύομαι, όνειρα μεγάλα. Αλλιώς θα ήμουν βουλευτή στο Σαμαρίνα, δεν είχα αυτή την προσέγγιση όταν ονειρεύεσαι στην Ευρώπη κάνεις μεγάλα όνειρα ελπίζοντας ότι κάνεις κάτι χρήσιμο. Γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την τροποποίηση και να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη μας πολιτικός και οικονομικός και οργανωτικός πιο κοντινή στον πολίτη, όχι μέσω ενός αναθεωρημένου ελληνικού κώδικα, αλλά και μέσω αλλαγής της δομής των τελωνίων. Ε, ώστε χώρες όπως η Ιταλία που έχουν διάφορα προβλήματα στις δομές τους να τις θέσουμε σε πιο σαφές, πιο καλό, πιο δημοκρατικό πλαίσιο. Εγώ αυτό περιμένω με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα προσπαθήσω να πετύχω με τη βοήθεια των συναδέλφων του Κοινοβουλίου για να καταλήξω σε μια πρόταση που θα ανοίξει ένα δρόμο επιτέλους πραγματικής εναρμόνισης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, θα δώσω το λόγο αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη, στον κύριο Τσιλιασκή. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε ευθύ αμέσως το λόγο. Πριν έρθω στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες που εκφράσατε, θέλω να σας πω ότι πράγματι το χρονοδιάγραμμα των Επιτροπών Ίντα και ΙΜΚΟ είναι πολύ σφιχτό. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι εσείς θέλετε να προχωρήσετε γρήγορα και σας είμαστε ευγνώμονες. Πρόκειται για την αναδιατύπωση. Συνεπώ δεν τροποποιούμε τίποτα στον ε, κορμό, στην ουσία. Έπρεπε όμως να αλλάξουν κάποια μικρά πραγματάκια γιατί χρειαζόντουσαν διευκρίνηση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τη στάση σας. Τώρα για τα ε, θέματα που θέσατε. Για τις ώρες. Υπάρχει το άρθρο 137, για το δείτε σε σχέση με το 135, Βλέπετε ότι εμεί θέλουμε την εναρμόνιση στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο, γιατί η εναρμόνιση των τελωνίων, των ορών εργασία των τελωνίων κτλ. είναι θέμα που είναι αρμοδιότητα και προνόμιο των χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, στο άρθρο 137, όπως σας είπα, προσπαθούμε να πετύχουμε αυτήν την εναρμόνιση όσο γίνεται περισσότερο. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει και αντικείμενο του τριμερούς διαλόγου, γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για μερικά, ίσως και πολλά κράτη-μέλη. Από την άλλη, προχωράμε στα ηλεκτρονικά τελωνία, ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλατε, αλλά πάντως αυτά θα είναι ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρο, τα ηλεκτρονικά δηλαδή τελωνιακά γραφεία. Ένα πολύ βέστητο θέμα είναι η εναρμόνιση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι τελωνιακοί κώδικες και τις ένωσεις προχωρούν. Εδώ, και πάλι σας είμαστε ευγνώμονες, έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παραμένουν όμως κάποιες αποκλήσεις της απόψης των χωρών μελών γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ διαφορετική κατάσταση από χώρα σε χώρα μεταξύ των 27. Προσπαθούμε όμως να την κάνουμε την εναρμόνιση ή όπου δεν γίνεται εναρμόνιση κάποια προσέγγιση. Πάντως φιλοδοξίες έχουμε και προσπαθούμε να εναρμονίζουμε ό,τι μπορούμε να εναρμονίσουμε. Για τον ΦΠΑ είναι φορολόγηση και το σύστημα πάλι διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και υπάρχουν ε, και οι διαδικασίες, 42 για παράδειγμα, και η ερμηνεία που δίνεται για τις ε, με καθυστέρηση επιστροφές. Και εδώ προσπαθούμε να έχουμε μια κάποια εναρμόνιση, αλλά το ΦΠΑ είναι πιο δύσκολο για την εναρμόνιση, γιατί παραμένει θέμα των ε, χωρών, παρόλο που έχουμε την οδηγία είναι προνόμιο και αρμοδιότητα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό των χωρών μελών. Αντίθετα με τον Τολυνιακό Κώδικα, από εκεί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Τέλος. Για την πληρωμή που γίνεται σε τρίτα μέρη. Είναι ένα εμπορικό ζήτημα και δεν μπορούμε άμεσα να παρέμβουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι πρέπει ε, γραπτά να δώσουμε μια απάντηση στην ερώτησή σας. Καταλαβαίνω ότι δεν σας ικανοποιεί αυτό που σας λέω τώρα, γι' αυτό και θα το κοιτάξουμε και θα σας απαντήσουμε γραπτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βασίζομαι στην απάντηση, θα μου στείλετε σύντομα. Είναι προφανές ότι κανένας από εμά δεν μπορεί να φανταστεί ότι μέσω αυτού του κανονισμού μπορεί να εναρμονίσει το ΦΠΑ. Αυτό όμως που ζητούμε είναι να εναρμονιστεί η μορφή των πληρωμών. Εξηγούμε. Είναι σαφές ότι στην Ιταλία μπορεί να βάλουμε το ΦΠΑ στο 30% και η Πορτογαλία να το βάλει στο 15% το ΦΠΑ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα που έχει κοινό φόρο, αυτό είναι δικαίωμα των κράτων μελών. Πιστεύω όμως ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι η απέτηση, η πληρωμή του ΦΠΑ, όπου, όποιο και να είναι το ποσοστό αυτού, θα πρέπει να γίνεται ίσπραξη με τον ίδιο τρόπο. Είτε εκτελονίζω στην Ολλανδία ή στη Γερμανία ή στην Τζένοβα, στην Ιταλία. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι κάποιες χώρες ε, ε, εισπράττουν ε, εισπράττουν μία-δύο φορές παραπάνω το, το ΦΠΑ ή επιστρέφουν με πιο αργούς χρόνους από ό,τι πρέπει. Άρα, δεν κάνουμε αυτό, μπαίνουμε σε πρόβλημα ανταγωνισμού. Διότι αν μια ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε την Ολλανδία, τυχαία, βάλει τη φορολόγηση ΦΠΑ τη χαμηλότερη όλων. Οπότε δουλεύουν τα τελωνία τις περισσότερες ώρες από όλα τα άλλα τελωνία και πώς να το πω τώρα και διευκολύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στο μέτρο του δυνατού είναι σαφές ότι όλοι εκείνοι που μπορούν θα επιλέξουν αυτά τα τελωνία για να φέρουν στην Ευρώπη εμπορεύματα. Συνεπώς, οι μεταφορείς αυτής της χώρας θα ωφεληθούν από δραστηριότητα, από δουλειά. Άρα, μέσω της δικής μας δουλειάς, των επομένων ημερών θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την πολιτική και οικονομική ένωση της Ευρώπης που αν δεν επιτεύχθη μέχρι τώρα μας οδηγεί σε καταστροφή. Αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τέσσερα πράγματα σε συνάρτηση με τη Λισαβόνα δεν θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους ναι, ούτε μας. Διότι εμείς χρονοτριβούμε και οι Ευρωπαίοι θα απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την Ευρώπη. Διότι με την κρίση τελευταία κανεί δεν μα θεωρεί πλέον αξιόπιστου. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά έτσι είναι. Εγώ λαμβάνω υπόψη αυτά που μας είπατε και αυτά που προτείνατε. Αν έχετε την καλοσύνη, λάβετε υπόψη και εσείς αυτά που λέω εγώ. Δηλαδή, ότι πρέπει να βρούμε ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει να προχωρήσουμε να μην καταλήξουμε στο Συμβούλιο με το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και για το κανονισμό για την ονομασία προέλευσης. Χρειαζόμαστε να φέρουμε μαζί μας ε, σίγουρα πράγματα και καλά για εκείνον που εργάζεται και παράγεται. Παράγει, συγγνώμη. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, υπενθυμίζω ότι στις 20, 29 Αυγούστου είναι η τελική προθεσμία γιατί 20 και 21 Ιουλίου θα έχουμε άλλη ανταλλαγή απόψεων, έτσι. Λοιπόν, 29 Αυγούστου είναι η τελική προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών 16 και 17-18 Σεπτεμβρίου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Εδώ βλέπω κάτι με το οποίο διαφωνώ. Πάμε στην Ολομέλεια του Απριλίου, λέει εδώ. Τι λέει. Απρίλη. Άρα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια. Διότι αν πάμε στην Επιτροπή τον Οκτώβριο και ο τριμερής διάλογος ξεκινά τον Φεβρουάριο, νομίζω ότι προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε να γίνει ο διάλογος το 2012. Έχω απογοητευτεί με την εμπειρία από τον κανονισμό για, την, ε, για τους κανόνες ε, προέλευσης, προστασίας προέλευσης κλπ. Οπότε θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τον Ιούλιο για να συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα. Οι επόμενε συνεδριάσει είναι 11 Ιουλίου από 9 με 12 και μισή και από τις 3 μέχρι τις 18 και 30 και στις 12 από τις 9 μέχρι τις 12 και 30 εδώ στις Βρυξέλλες προφανώς. Ευτυχώς ολοκληρώσαμε το μεταξύ αυτή τη μακρά σύνοδο ψηφοφοριών. Ευχαριστώ τους ελάχιστους παρόντες που υπήρξαν αλληλέγγυοι μέχρι τέρμα μέχρι τέλους και θα τα ξαναπούμε τον Ιούλιο. Γεια σας και καλή όρεξη.